chiedo ai colleghi di prendere posto così possiamo proseguire. Συνεχίσουμε λοιπόν με τις προσπάθειές μας. Θα δώσω το λόγο στην Φεντερίκα Μογκερίνη, την είπατε εκπρόσωπο για εξωτερικά θέματα, να σας ενημερώσω ότι δεν έχει τεθεί, να ζητηθεί μάλλον να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 4 του κανονισμού και γι' αυτό μια τέτοια αλλαγή η οποία προτάθηκε θεωρείται δεκτή. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα στην ημερήσια διάταξη, δηλώσεις της Αντιπροέδρου, είπα της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης